Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να αρχίσουμε. Ich begrüße Sie Σας χαιρετίζω όλους στην, πιο σύντομη, λίγο πιο σύντομη συνεδρίασή μας σήμερα. Αλλά πιστεύω πως το χρόνο που έχουμε θα τα καταφέρουμε καλά, αν και έχουμε κάποιες εκτενείς ψηφοφορίες Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν συμφωνείτε με το σχέδιο της ημερησίας διάταξης, με την μορφή που έχει ή αν υπάρχουν επιθυμίες συμπλήρωσης ή τροποποίησης της ίδιας. Δεν συντρέχει αυτό, οπότε εγκρίνεται η ημερησία διάταξη όπως έχει. Σημείο 2, ανακοινώσεις του Προέδρου. Θα ήθελα να σας ενημερώσω πως σήμερα έχουμε στις εξής γλώσσες διερμηνία γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, τσεχικά, εσθονικά, ουγγαρικά, πολωνικά, βουλγαρικά και ρουμανικά. Εκτός αυτού, πρέπει να σας υποδείξω πως όπως πάντα γίνεται αναμετάδοση της συνεδρίασης στο διαδίκτυο. Οι αποφάσεις των συντονιστών της 25ης Απριλίου σας απεστάλησαν στις 28 Απριλίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όπως πάντα πιστεύω πώς μπορούμε να θεωρήσουμε τα πρακτικά ως εγκεκριμένα, καθώς έως την προθεσμία της 3ης Μαΐου δεν υπήρξαν κάποιες ενστάσεις από πλευρά σας. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Έχουμε ψηφοφορίες επί τριών γνωμοδοτήσεων και θα ήθελα να αρχίσω κατευθείαν με την πρώτη. Είναι η γνωμοδότηση σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ελεκτρονικών Επικοινωνιών ο Κούρτσιο Μαλτέζα ήταν ο εισηγητή μου. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Κούρτσιο αν θέλει να λάβει σύντομα το λόγο. Εντάξει. Οπότε περνάμε στην ψηφοφορία και αρχίζουμε με την τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 τροπολογία 89 κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία για να δούμε μέχρι να βρει ο Σίλβιο την κάρτα του οπότε κηρύσω το πέρας της ψηφοφορίας. Δώδεκα προς 8 εγκρίνεται. Περνούμε στο δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. 90. Τροπολογία 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 και 91. Ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επαλήθευση. Εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 11 προς 10 ψήφι εγκρίνεται. Τροπολογία 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 97 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πάμε στην τροπολογία 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Πάμε στην τροπολογία 98. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως εγκρίνεται, αλλά θα ήθελα να το επαληθεύσω. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 13 προς 9 εγκρίνεται. Τροπολογία 101 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 102 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 και 104 υπέρ 18 και 104 Η 104 έχει αποσυρθεί αλλά η 18 υπάρχει ακόμα 18 υπέρ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 κατά αποχές απορρίπτεται 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συγγνώμη νομίζω απορρίφθηκε λάθος δικό μου θα το επαληθεύσουμε όμως 23 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ναι, σαφώς και απορρίπτεται, συγγνώμη, λάθος δικό μου. Τροπολογία 110 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 και 123 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αυτό θα ήθελα να το επαληθεύσω. 25 άρχεται η ψηφοφορία Τώρα πρέπει να κηρύξω το πέρας της ψηφοφορίας. Πέρας. Με 13 προς 12 εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να το απελευθεύσουμε. Ας το απελευθεύσουμε λοιπόν. 27 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 14 προς 10 εγκρίνεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 όχι 28 καταπίπτει 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές νομίζω πως απορρίπτεται αλλά θα ήθελα να το επαληθεύσω 127 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ναι, απορρίπτεται, λάθος έκανα. 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ας το επαληθεύσουμε αλλά νομίζω πως ήταν σαφές άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεν ήταν τόσο σαφές το αποτέλεσμα 13 προς 12 αλλά δίκιο είχα εγκρίνεται συγγνώμη συγγνώμη μου έμοιαζε πιο σαφής η κατάσταση. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 131 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 17 προς 6, συγγνώμη λάθος δικό μου. Θα παρακαλούσα να μου το δείχνετε σαφώς, ώστε να έχω μια καλύτερη εικόνα από εδώ. 132. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 133 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές πολύ, πάλι οριακό το αποτέλεσμα επαλήθευση 135 άρχεται η ψηφοφορία πέρας 11 προς 14 απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οπότε επαναλαμβάνουμε υπέρ, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να το επαληθεύσουμε επειδή είναι οριακό το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 13 προς 13 απορρίπτεται 137 υπέρ απορρίφθηκε ούτως ή άλλως θα ήταν 14 προς 13 τότε 14 προς 13 τότε. 137 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ κατά αποχές ε, ε, απορρίπτεται 146 υπέρ κατά αποχές αυτό πρέπει να το ελέγξουμε 146 άρχεται η ψηφοφορία πέρας 13 προς 14 απορρίπτεται ναι η Τζούλη έχει την κάρτα της 13 προς 14 απορρίπτεται 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές θα ήθελα να το επαληθεύσω Άρχεται ψηφοφορία για την 33. Πέρας. Ένα μέλος του SND παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Τώρα είμαστε εντάξει. Πέρας. 13 προς 14. Απορρίπτεται. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω πως απορρίπτεται αλλά και αυτό θα ήθελα να το επαληθεύσω. 149 λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 11 προς 14 απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ κατά αποχές και εδώ θα ήθελα να προβώ επαλήθευση 151 άρχεται η ψηφοφορία πέρας 14 προς 13 εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 153 υπέρ κατά αποχές νομίζω πως εγκρίνεται αλλά και αυτό θα ήθελα να το επαληθεύσω άρχεται η ψηφοφορία 153 πέρας 16 προς 11 εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συγγνώμη 36 καταπίπτει 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές θα ήθελα να το επαληθεύσω επειδή υπήρξαν κάποιες αποχές, δεν είμαι σίγουρη. Άρχεται η ψηφοφορία για την 154. Πέρας. 12 προς 10 εγκρίνεται με 5 αποχές. 155 υπέρ κατά αποχές Εάν το S&D σήκωνε τα χεράκια του, αυτό θα με βοηθούσε πολύ. 155 υπέρ, άλλη μια φορά. Κατά. Αποχές. Πάλι δεν έχω καλύτερη εικόνα. Επαλήθευση λοιπόν. 155. Λυπάμαι. Πέρας. 10 προς 16 απορρίπτεται. 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές σαφώς εγκρίνεται ένα σαφές αποτέλεσμα 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 162 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ 40 κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές θα ήθελα να την επαληθεύσω άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 2 3 συγγνώμη επί της τροπολογίας 3 πέρας 17, 10 προς 17 απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ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 Ναι, δίκιο έχετε, είπα το 54 δύο φορές, 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 και 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές θα ήθελα να το επαληθεύσω άρχεται η ψηφοφορία πέρας 13 προς 15 απορρίπτεται 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίπτεται αλλά να το επαληθεύσουμε 88 άρχεται η ψηφοφορία πέρας 15 προς 13 εγκρίνεται Πάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. 24 υπέρ, 0 κατά, 4 αποχές. Η έκθεση εγκρίνεται ως έχει. Να συγχαρώ τον εισηγητή. Περνάμε τώρα στη γνωμοδότηση για τον φορέα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η Σίλβια Κώστα τα εισηγήτρια. Θέλεις να πεις κάτι? Λοιπόν, Μπέρεκ. Σίλβια, θέλεις να πεις κάτι? Θέλω να ευχαριστήσω τους και όλους και την γραμματεία ε, όλους τους ε, βοηθούς, το προσωπικό. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποια επίμαχα ζητήματα, ε, όμως ε, γνωρίζω ότι η Επιτροπή θέλει να κάνει το βήμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στην ψηφοφορία 20 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 56 και 57 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ήθελα να το παληθεύσω. 56 και 57 άρχεται η ψηφοφορία. Geschlossen. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η ισοψηφία. 55 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική πρόταση παρελθόν 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στη συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κα, υπε, κατά ζητώ συγγνώμη 68 68 και 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνονται εγκρίνεται 72 και 74 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 και 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ 79, συγγνώμη, 79 λέει η πρόεδρος, διορθώνει. 79 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 81 και 82 υπέρ, κατά, αποχές, επιβεβαιώνουμε ηλεκτρονικά. 81 και 82 ψηφίζουμε. Λήξη πληροφορία. Απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 86 και 87 υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι η κατάσταση είναι όπως πριν, οπότε θα απορριφθεί, αλλά α επιβεβαιώσουμε ηλεκτρονικά. 86-87, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Geschlossen. Λήξη ψηφοφορία. Αντίστροφα αυτή τη φορά. 15 υπέρ, 13 κατά. 89 και 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και εδώ θέλω ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ένα ψηφοφορίας. Geschlossen. Λήξη ψηφοφορίας. 15 κατά 13 υπέρ απορρίπτεται. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονική επαλήθευση αφού το ζητάτε 94 άρχεται η ψηφοφορία λήξη ψηφοφορίας 16 υπέρ 12 κατά εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται α, ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία λήξη ψηφοφορίας 16 κατά 11 υπέρ απορρίπτεται 97 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά εποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά σε επαληθεύσουμε. Λήξη ψηφοφορία 15 κατά 13 υπέρ απορρίπτεται. 100 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 102 υπέρ κατά εποχές Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Για την 102. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορία. Ισοψηφία. Άρα απορρίπτεται. 103 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 127 και 128 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Δεκαπέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά Εποχέ. απορρίπτεται 3 συμβαστική πρόταση 3 υπέρ κατά Εποχέ. υπέρ εγκρίνεται ενώ 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στην 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική πρόταση παριθμών 5 υπέρ κατά Εγκρίνεται η 12 υπέρ κατά Εποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 12 άρχεται. Λίγη ψηφοφορία. 17 κατά, 11 υπέρ, απορρίπτεται. 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 122 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση παριθμών 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για την 134 άρχεται λίγη 11 υπέρ 17 κατά απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση Έλξη ψηφοφορία 22 υπέρ 6 κατά Εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη, δεν εκτιμώ σωστά την κατάσταση γιατί δεν καταλάβαμε πολύ καλά τα χέρια. 137 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική παριθμόν 7 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 140 υπέρ. Κατά. Α, απορρίπτεται 141 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται να το απαληθεύσουμε. για την 141 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά κλείνει η ψηφοφορία 12 υπέρ 16 κατά απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά εποχέ. απορρίπτεται 24 υπέρ κατά Κατά, ε, απορρίπτεται 1 υπέρ κατά εποχέ. εγκρίνεται 25 υπέρ κατά εποχέ. εγκρίνεται η ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 25 εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ 3 ε, κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 ε, α, επαλήθευση Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 5. 13 υπέρ, δεκαπέντε κατά. Απορρίπτεται. Ζητώ συγγνώμη. 36 υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ όχι 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 όχι ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 42 43 λέει η πρόεδρος λίγη ισοφορία Α, 42 42 διορθώνει η πρόεδρος 13 υπέρ 15 κατά απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές Τι σημαίνει με το ΕΛΚ. Όχι, ε, δεν τη δέχεστε. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου. Η ε, ηλεκτρονική σουφορία, άρχεται. Λίγη σουφορία. 15 υπέρ, 13 κατά. Εγκρίνεται. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν οριακό. Συγγνώμη για τις πολλές επαληθέσεις, αλλά χρειάζονταν. Οπότε περνούμε στην τελευταία ψηφοφορία της σημερινής μέρας. Είναι η γνωμοδότηση της συναδέλφου Λυριάντα σχετικά με την ευρωπαϊκή δράση για τη βιωσιμότητα. Είναι εδώ η συγκήτρια. Ναι, παρακαλώ, θα θέλατε το λόγο, ορίστε. Ναι, πολύ σύντομα. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τους σκιώδεις και τη γραμματεία για τις συστάσεις και τη βοήθεια που προσέφεραν. Οι γνωμοδοτήσεις, όπως ξέρουμε, πρέπει να είναι σύντομες και έβλητες. Όταν τις συντάξαμε, αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε στην, στο στόχο SDG 4 ε, από το σχετικό πλαίσιο θα ήθελα να έχει ευρύτερο πεδίο η γνωμοδότηση δική μου, αλλά δεν το επέτρεπαν οι χαρακτήρες και τα όρια. Γι' αυτό ε, προσπέθησα να επικεντρωθούν στο κεντρικό στόχο που είχαμε θέσει. Το γεγονό ότι το 2010 2014 οι επενδύσει στην εκπαίδευση και την κατάρταση αυξήθηκαν κατά 2,5%. Γνωρίζουμε πολύ καλά όμω ότι με το Brexit εν ώψη αυτό δεν θα βελτιωθεί, οπότε πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή και πρέπει να δείξουμε πυγμή και να προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε τουλάχιστον αυτέ τι γραμμέ που είναι τόσο σημαντικέ για την ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.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 αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε στην τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Εάν εγκριθεί το πρώτο τμήμα, απορριφθεί μάλλον, τότε καταπίπτει το δεύτερο τμήμα. Τώρα ψηφοφορία για το πρώτο, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές θα το επαληθεύσουμε επειδή είδα μόνο πολύ λίγα χεράκια. Δεύτερο τμήμα της 31 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας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 Καθώς δεν έχουμε πολύ χρόνο και οι ψηφοφορίες σαν λίγο περισσότερο από ό,τι σχεδιάσαμε, θα ήθελα να προχωρήσω με την μυρίσια διάταξη, για την οποία έχουμε μόνο κάτι περισσότερο από μισή ώρα, επειδή στη συνέχεια έχουμε αμέσως τη συνεδρίαση των συντονιστών. Γι' αυτό και θα παρακαλούσα να έχουμε συγκεντρωμένες διαβουλεύσεις. Περνούμε στο σημείο 6, εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης. Παρακαλώ, αποχωρήστε ήσυχα. Εάν θέλετε να μιλήσετε, να συζητήσετε, παρακαλούμε αποχωρήστε και αφήστε μας να εργαστούμε εδώ. Λοιπόν, εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης για την έκθεση είναι της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής προνογραφίας. Είναι και για μας ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ήδη κατά την τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο ασχοληθήκαμε πολύ διεξοδικά με το θέμα και επίσης καταθέσαμε μια σχετική γνωμοδότηση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Στην περίπτωση της σεξουαλικής κακοποίησης πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρές αξιόπινες πράξεις για την καταπολέμηση των οποίων χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση. Και αυτό ήδη το Δεκέμβριο του 2011 το τονίσαμε στην οδηγία που εγκρίθηκε. Η συγκίτριά μας είναι η Ζαμπίνε Φερχάιεν. Στη συνέχεια θα ήθελα να δώσω τον λόγο στους Σκιώδης και σε άλλα μέλη, εάν επιθυμούν να πάρουν το λόγο. Και στο τέλος θα ήθελα να πάρω και εγώ το λόγο. Παρακαλώ πρώτα η Ζαμπίνε Φερχάιεν να μας παρουσιάσει σύντομα την έκθεσή της. Ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση ασχολείται με το ότι στην τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο εγκρίναμε ένα νομικό κείμενο για την προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και στο διαδίκτυο διευρύναμε το θέμα, υπήρξαν κάποιες αξιόπινες πράξεις όπως το grooming που επίσης ορίστηκαν ως αξιόπινες πράξεις. Τώρα από την έκθεση εφαρμογής, δηλαδή κατά πόσον μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών οι αλλαγές αυτές. Εδώ βλέπουμε μια διαφορετική πυκνότητα μεταφοράς, ιδίως όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, δηλαδή τα μη νομοθετικά μέτρα, αλλά επίσης τη φροντίδα, τη μέρημνα για τα θύματα Εκεί ακόμα κάποια πράγματα παραμένουν αόριστα και εδώ πιστεύω πως πρέπει να υποδείξουμε στα κράτη-μέλη πως πρέπει να προβούν σε σχετικές δράσεις. Επίσης λόγω των τεχνικών εξελίξεων στο διαδίκτυο όσον αφορά τις τεχνολογίες κωδικοποίησης, το σκοτεινό διαδίκτυο, έχουμε φτάσει στο σημείο όλο και περισσότερο από το ανοιχτό διαδίκτυο να μπορεί κανείς να μπει στο λεγόμενο βαθύ διαδίκτυο ή να έχουν μετατεθεί τέτοια περιεχόμενα στο σκοτεινό διαδίκτυο, οπότε είναι όλο και πιο δύσκολη η ποινική δίωξη. Διαφέρουν οι απόψει μα όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα. Υπάρχουν διάφορε μορφέ. Αφενό, ο αποκλεισμό ή η διαγραφή, εκεί σημειώθηκε μεγάλη πρόοδο όσον αφορά το συντονισμό, ιδίω και τι διαδικασίε διαγραφή μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών μελών αλλά δεν αρκούν οι προσπάθειέ μας σε όλου του τομεί, ιδίω αν πρόκειται για τομεί οι οποίοι δεν είναι προσβάσιμοι στο ανοιχτό διαδίκτυο, αλλά κρύβονται στο λεγόμενο βαθύ διαδίκτυο ή σκοτεινό διαδίκτυο, ανάλογα με τον όρο που επιλέγει κανεί, αν και το σκοτεινό διαδίκτυο δεν εκπροσωπεί παρά μια συγκεκριμένη τεχνολογία. Εκεί επιθυμούμε μια πιο αυστηρή ποινική δίωξη και καλύτερο συντονισμό όταν το αντικείμενο δεν είναι μόνο το υλικό σεξουαλικής κακοποίηση, αλλά επίσης για την κακοποίηση κάθε αυτή στην πραγματικότητα. Δηλαδή την εμπορία παιδιών είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό και με την έκθεσή μας αυτή θέλουμε να προτρέψουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν, να μεταφέρουν κατάλληλα τις νομικές διατάξεις που εγκρίναμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο εσωτερικό του δίκαιο και επιτέλους να ταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο. Πιστεύω πως τα παιδιά είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Οι παιδικές ψυχές και τα παιδικά σώματα εκτίθενται σε τέτοιες πράξεις και καταστρέφονται από τέτοιες πράξεις, το οποίο είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορούμε να ανεχτούμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή αυτή. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους σκιώδες εισηγητές. Πρώτον, πρώτη η κυρία Μέτσικ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η κυρία Φερχάιρεν έχει συντάξει μια πολύ καλή και ισόρροπη νομοδότηση. Με πάρα πολύ εύστοχες προτάσεις, οι οποίες πραγματικά ε, καλύπτουν τα βασικά σημεία της οδηγίας για την ε, σεξουαλική κακοποίηση και την εκμετάλλευση των παιδιών και την παιδική πορνογραφία. Από αυτή λοιπόν τη σκοπιά νομίζω ότι είναι πολύ ε, σωστά ισορροπημένη έκθεση. Επίσης χαίρομαι που η συγγετρία επικεντρώνεται στις βασικές προτεραιότητες και όλος ιδιαίτερος στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση, καθώς και την κατάρτιση και εκπαίδευση και την υποστήριξη των θυμάτων, την ε, διερεύνηση των ε, εγκληματικών ενεργειών και την δίωξη των δραστών. Είναι πολύ καλή ε, αντίδραση, κοκτέιλ αντίδραση, για να το πω έτσι, σε αυτή τη μάστιγα του 20ου αιώνα. Ε, αυτοί που δεν διστάζουν να ε, προβάλλουν τα παιδιά του στο διαδίκτυο θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερω. Και γι' αυτό έχω κάνει μια σειρά από προτάσει με τι τροπολογίε μου. Πρώτα απ' όλα την πρόληψη. Θα πρέπει να υπάρξει ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και παραδειγμάτων. Εδώ θα προσπαθήσω να μην συνοπτική λόγω περιορισμού χρόνου. Επίση, τα νέα κυβερνοεγκλήματα όπως η ειδονοβλεψία και η αντεστραμμένη πορνογραφία. Επίσης, η εκπαίδευση και η κατάρτιση και για τα παιδιά και για τους ενηλίκους, ιδίως για τους γονείς και όλους όσοι έρχονται σε επαφή με τα παιδιά θα ήθελα να υποστηρίξω την, ε, το όριο ηλικία για να μπορεί κανεί να χρησιμοποιεί εργαλεία ανάλογα από την ηλικία του και να προωθηθεί ο αλφαβητισμός, ε, η γνώση δηλαδή των ε, ηλεκτρονικών μέσων ανάλογα με την ηλικία. Επίση, η προστασία των παιδιών να τα φτάνουν στα δικαστήρια, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών. Και αυτό κάποιε φορέ εξαρτάται από του ενηλίκου και του γονεί συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ζωτικής ε, σημασίας για να εντοπιστεί και να καταπολεμηθεί το παράνομο περιεχόμενο αλλά και να διωχθεί ο κάθε υπεύθυνο για την επιγραμμική του ε, ανάρτηση. Επίσης, η σεξουαλική κακοποίηση επιγραμμικός στο διαδίκτυο καθώς και υποβολή εκθέσεων με τρόπο ασφαλή και ε, διαρθρωμένο για τα παιδιά και προστασία των θυμάτων. Επίσης, ευξανόμενη απειλή για τα παιδιά που πλήττονται από την κρίση των προσφύγων ε, είναι εκτεθειμένα σε σεξουαλική κακοποίηση και ε, κάποιες φορές σε εκμετάλλευση. Επίσης τα ε, ιδιαίτερα δίκτυα, τα παράνομα δίκτυα που έχουν παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να αποσύρεται, αλλά αυτό να γίνεται βάση σαφών και διαφανών κριτηρίων που να παράσχουν τα ε, ανάλογα επίπεδα νομικής βεβαιότητας και να συμμορφωνόνται με τι ισχύουσε νομικέ και δικαστικέ διαδικασίε. Υποστηρίζω πλήρω λοιπόν την εισηγήτρια σε αυτή την άριστη εκθεσή τη και ανυπομονώ για τη συνεργασία με τους υπόλοιπους κοιόδης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έμα Μακλάρκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρου του ECR, στη συνεργασία με τους συναδέλφους, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δώσουμε στα κρατημέλη τη δυνατότητα να συνεργαστούν και να μοιραστούν τις καλύτερες πρακτικές για την εξάλληψη της σεξουαλικής κακοποίηση πρόκειται για διασυνοριακά εγκλήματα και πρέπει να δείξουμε πως προστατεύουμε τα παιδιά και πρέπει να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Οι τεχνολογικές εξελίξεις τις τελευταίες δεκαετίες αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέστησαν πιο εύκολη και πιο γρήγορη την πρόσβαση σε τέτοιο υλικό και δυστυχώς επίσης διευκόλυναν την διάδοση τέτοιου υλικού από εγκληματίες. Γι' αυτό και οι πολιτικοί εργάζονται συνεχώς για την ε, δημιουργία εναλλακτικών για την αποτροπή του φαινομένου αυτού. Και αυτό μας δίνει την ευκαιρία ως Επιτροπή να προτείνουμε κάποιες ξεκάθαρες κατευθυντηρίες γραμμές για τα κράτη-μέλη, αλλά επίσης για να προτείνουμε ευκαιρίες βελτίωσης είναι δύο σημεία για τα κράτη-μέλη. Το πρώτο από αφορά τη διακίνηση τέτοιου υλικού και το δεύτερο τη διασπάληση φραγμών. Όπως λέει ξεκάθαρα η οδηγία, τα κράτη-μέλη πρέπει να ακολουθήσουν το σαφές παράδειγμα του Internet Watch Foundation στο Ηνωμένο Βασίλειο και πρέπει να ενεργοποιήσουν ανοιχτές γραμμές επικοινωνίες για τον εντοπισμό υλικού παιδικής κακοποίησης. Έτσι, λόγω αυτής της πολιτικής μηδενικής ανοχής, επιτύχαμε δραματική μείωση του φαινομένου. Πρέπει να δείξουμε πως αυτοί που διαπράττουν τέτοια εγκλήματα έχουν να αντιμετωπίσουν την σκληρότατη δίωξη στα κράτη-μέλη Πρέπει να δείξουμε πως εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη-μέλη έχουμε μια ξεκάθαρη γραμμή και συνεργαζόμαστε με άλλα έθνη ανά τον κόσμο για να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ πολύ. Η, σκιο... η συγγήτρια των Πρασίνων δεν είναι εδώ. Χέλγα, θα ήθελες... Ε, Ευχαριστώ και εγώ βλέπω ένα μεγάλο πρόβλημα με το ανοιχτό διαδίκτυο και το σκοτεινό διαδίκτυο ό,τι αφορά την ε, κακή αντίληψη και ε, συμπερίληψη των παιδιών. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτά που συμβαίνουν και τα διάφορα φαινόμενα που περιγράφουμε διαρκώς επιδεινώνονται. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αυτή τη διαφωνία που μπορεί να υπάρχει μεταξύ ελευθερία της έκφρασης από τη μια και από την άλλη την προστασία και πρόληψη της ε, κακής ε, συμπερίληψης και χρήσης, για να το πάει στον των παιδιών στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφή κριτήρια για το περιεχόμενο που μπορεί να περιλαμβάνεται στο διαδίκτυο και να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις. Αυτή είναι η βασική μέρημνα που θέλω να καταστεί σαφής και να μας οδηγήσει και αυτό το κάνουν όχι μόνο οι ιδιωτικές εταιρείες. Ε, ό,τι δεν συμφωνεί με, το μηχανισμό να μπορεί να ε, εντοπίζεται και να υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση για να έχουμε τη σωστή αντιδράση. Δεν μπορεί να παραβιάζονται οι αρχές του κράτους δικαίου και της νομικής βεβαιότητας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Έμπλεξα λίγο τη σειρά. Κανονικά με τη σειρά των πολιτικών ομάδων πρώτα θα είχε σειρά η Άλντε. Ο Σκιώδης ωστόσο δεν βρίσκεται εδώ. Γι' αυτό και θα δώσω τον λόγο στη Μαρτίνα Μίχελς. Ναι, έχουμε μια αλλαγή στη σειρά. Θα ήθελα να συνεχίσω σε αυτό που είπε η κυρία Τρούπελ μόλις πως το πρόβλημα εδώ είναι η ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας της έκφρασης και του κράτους δικαίου. Πολλά από αυτά που υπόθηκαν δεν είναι νέα. Αλλά αν λύσουμε όλα τα επιμέρους προβλήματα, πάντα καταλήγουμε στο βασικό πρόβλημα, ότι δηλαδή οι αξιόπινες πράξεις και τα υλικά αυτά διαδίδονται πολύ εύκολα στο διαδίκτυο, αλλά δεν δημιουργούνται στο διαδίκτυο, δημιουργούνται πιο πριν. Γι' αυτό και είναι το ερώτημα πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε το πρόβλημα αυτό. Δηλαδή την παραγωγή φωτογραφιών και την εκμετάλλευση παιδιών, δηλαδή πώς μπορούμε να δράσουμε περισσότερο προληπτικά. Και πιστεύω πως κάθισετε σαφές πως και αρκετά χρόνια μετά από την οδηγία αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες όσον αφορά το διαδίκτυο και εγώ θα ήθελα να πω πως είμαι πεπισμένη πως η αρχή της διαγραφής αντί του αποκλεισμού έως σήμερα τουλάχιστον για μένα είναι η μόνη διαδικασία με νόημα ενάντια σε αυτές τις παράνομες εικόνες και τα παράνομα βίντεο όπως και η δίωξη της παιδικής πορνογραφίας εκτός διαδικτύου. Η παιδική πορνογραφία είναι δύσκολο να καταπολεμηθεί μέσω φραγμών στο διαδίκτυο, αποκλεισμών στο διαδίκτυο, καθώς οι αποκλεισμοί δεν βοηθούν, δεν έχουν αποτέλεσμα για την τέλεση της αξιόπινης πράξης. Και παρά τα όσα προτείνουμε, ούτε κατά προσέγγιση μέσω γενικών διατυπώσεων δεν κατορθώνουμε να φτάσουμε την κατεύθυνση να ταχθούμε υπέρ του αποκλεισμού. Η οδηγία του 2011 τάσεται ξεκάθαρα υπέρ της διαγραφής και πιστεύω πως αυτό πρέπει να το προσυπογράψουμε και να το εξειδικεύσουμε. Με τη γνωμοδότηση επίσης άρχισε και πάλι η συζήτηση για την ευθύνη για τα περιεχόμενα από τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου. Ας ρωτήσουμε για την ευθύνη των πλατφορμών κοινής χρήσης βίντεο διαδίδουν οπτικοακουστικό υλικό ακόμη και αν το ορίσουμε με την συγκεκριμένη οδηγία. Το είπε ήδη η προλαλή σα από το S&D. Χρειαζόμαστε περισσότερα προγράμματα για τη βελτίωση του αλφαβητισμού στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, κυρίως για γονείς και εκπαιδευτικό προσωπικό. Πιστεύω πως αυτό είναι εξίσου σημαντικό όσο οι τεχνικές λύσεις. Σε γενικές γραμμές πιστεύω πως συμφωνούμε με την εισηγήτρια την οποία και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ από τους σκιώδεις εισηγητές δεν είναι κάποιος εδώ γι' αυτό και περνώ στου, στα υπόλοιπα μέλη παρακαλώ περιοριστείτε στο ένα λεπτό Ζούλη Γουότ πρώτη uh, yes, I... Ναι, απλώς να πω αυτό που είπε και η Έμα Μακλάρκιν ο καλύτερος τρόπος να προστατεύσουμε τα παιδιά ως ευάλωτα πρόσωπα είναι να συνεργαστούμε διασυνοριακά. Αυτό ακριβώ είναι σχεδιασμένο να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το βρίσκω εξαιρετικά υποκριτικό να λέει η κυρία Μακλάρκιν σε αυτή την επιτροπή, επειδή είναι υπέρ του Brexit, να θέτει ένα αμφιβόλο την ασφάλεια των ε, παιδιών και των νεαρών ανθρώπων, όχι μόνο στον Ηνωμένο αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Εγώ εργάστηκα με παιδιά και νέου ανθρώπου που είναι ευάλωτα. Έχω εργαστεί με τι ενώσει και τα κέντρα που φροντίζουν για την ασφάλεια των παιδιών και γνωρίζω πολύ καλά καλά ότι ανησυχούν ιδιαίτερω για τον αντίκτυπο του Brexit στα πλέον ευάλωτα άτομα του πληθυσμού. Θέλω λοιπόν να καταγγείλω την υποκριτική στάση αυτής της βουλευτού που είναι υπέρ του Brexit. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γραμματικάκης. Ε, εγώ θα είμαι πολύ σύντομος ε, κύριε Πρόεδρε. Ο συνήθως Νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η εισήγηση, η προσπάθεια. Έχω όμως μια εντύπωση ότι πάντα είμαστε λίγο πίσω, χωρίς να φταίμε εμείς, από τις εξελίξεις. Δηλαδή, ας το πω, η κακοποιή του διαδικτύου είναι πολύ πιο αποφασισμένη και είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από μας. Και θα ήθελα εκεί να δώσουμε την προσοχή μας, δηλαδή στην πρόληψη, να είμαστε εμείς μπροστά να σταματάμε τις προσπάθειές τους και δεύτερον να υπογραμμίσω ένα πολύ σημαντικό σημείο που ακούστηκε εδώ είναι οι πληροφορίες, οι έγκυρες πληροφορίες, οι μελέτες ότι παρόμοια περιστατικά απεχθεί εξασκώνται στα παιδιά των προσφύγων. Το προσφυγικό θέμα είναι τεράστιο, το ξέρετε όλοι, το ξέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ιδιαίτερα για τα παιδιά είναι ένα φαινόμενο εγκληματικό και νομίζω θα πρέπει η εισήγησή μας να δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, Σιλβία Κώστα. Εκτίμησα ιδιαίτερα την γνωμοδότηση της Σαμπίν Φερχάριν, διότι αγγίζει δύο πτυχές. Αυτή που πιο πολύ αφορά την Επιτροπή μας, διότι ίσως ε, στα θέματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στην σχετική έκθεση δεν υπάρχουν τόσα πολλά. Πρέπει να επικεντρωθούμε δηλαδή στο σκέλος που αφορά την διοργάνωση και τη συνεργασία των διεθνών και των εθνικών συστημάτων. Είναι πολύ σημαντικό πάντως να ε, θυμίζουμε τι γίνεται ε, με το διαδίκτυο, με τα τηλεφωνικά δίκτυα που αυτή τη στιγμή λειτουργούν ε, σε 44 χώρες σε συνεργασία και όπως το WhatsApp και να δούμε και θέματα πιο ευαίσθητα, όπως πώς θα παρέμβουμε για να ειδοποιούμε για ποινικέ αξιόπινε πράξει ή εγκλήματα που γίνονται εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτό τη δική μα επικράτεια. Το άλλο θέμα είναι πώ θα δώσουμε έμφαση στην εκπαίδευση ακριβώς των ε, ε, διαχειριστών του όλου συστήματος και των φορέων. Των φορέων στο σχολείο, στη δικαιοσύνη όλων ε, όσων όσοι συμμετέχουν στην και έχουν επαφή με τα παιδιά. Οι μισές περίπου, ίσως και παραπάνω χώρες, ενέκριναν ομαδικά αυτή τον κανόνα με τα διάφορα site που πρέπει να μπλοκάρονται. Εδώ Μιλάμε για 72 ώρες κατά μέσο όρο για να μπορέσει κανείς να ζητήσει την απόσυρση του περιεχομένου από συγκεκριμένα δίκτυα. Εδώ υπήρξαν ε, προβλήματα με ανηλίκους πολλές φορές στην Ιταλία λόγω αυτού του κανόνα. Ευχαριστώ πολύ. Έμα Μακλάκεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να επανέλθω στα σχόλια της κυρίας Ward ε, από εκεί. Το βρίσκω πραγματικά πίστευτο που κάποιος χρησιμοποιεί σε μια τέτοια συζήτηση τόσο σημαντική τις πολιτικές του απόψεις και σκοπιμότητες. Είναι κάτι που αναγνωρίζουμε πλήρως. Δεν έχει σύνορα αυτό το έγκλημα. Είναι έγκλημα διεθνούς χαρακτήρα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε από κενού. Και βεβαίως το Ενωμένο Βασίλειο εδώ έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε όλο τον κόσμο. Δεν πρέπει να σταματήσουμε το πρόβλημα επικεντρωνόμενοι στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Πρέπει να συνεργαστούμε διεθνώς. Δηλαδή τι, δεν θα ε, συνεργαστούμε με τον Καναδά ή δεν θα δούμε ε, τι γίνεται αλλού. Τα σύνορά μας μετακινούνται, μεγαλώνουν. Ε, πρέπει να κινηθούμε και εμείς προς την ίδια κατεύθυνση Εργάζομαι με το θέμα του εδώ και πολλά χρόνια και θα συνεχίσω να κάνω το ίδιο όσο είμαστε πλήρη μέλη τη Ένωση αυτή, αλλά το ίδιο και όταν φύγουμε. Το ίδιο. Διότι είναι θεμελιώδου σημασία για την ασφάλεια και την προστασία των νεών γενεών. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και θα έπρεπε όλοι να οδεύουν προ την ίδια κατεύθυνση. Και τώρα και μετά τον Brexit. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω πως τώρα δεν πρέπει να συζητήσουμε για το Brexit αλλά να συγκεντρωθούμε στο θέμα. Τώρα θα ζητήσω, θα ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν έχει κάποιες παρατηρήσεις. Υπάρχει ένας εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ορίστε το πολύ δύο λεπτά παρακαλώ, αν γίνεται. Thank you very much, uh, Madam uh, Chair. And... Uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε και την Επιτροπή σας που συντάξετε αυτή την έκθεση. Η Επιτροπή καλωσορίζει την ομοδότηση τονίζει κάποια από τα κύρια ζητήματα που το χειριζόμαστε στην καθημερινή μας δουλειά για την καταπολέμηση της ε, παιδικής, ε, της εκμετάλλευσης και της ε, κακοποίησης των παιδιών εκτός και εντός διαδικτύου. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση τη Επιτροπή από το Δεκέμβριο πέρσι και στην μεταφορά από τα διάφορα κράτη περιμένουμε να ε, ε, μεταφέρουν σωστά την οδηγία του 2011. Και αυτό το σχέδιο χρηματοδότηση χρησιμοποιεί κάποια από τα ζητήματα που έχουν ε, ανακύψει και τα έχουμε εντοπίσει και εμεί όχι απαραίτητο συμπεριλάβει στην οδηγία, αλλά έχουμε αρχίσει να τα μελετούμε. Ήθελα να τονίσω τρία από αυτά, όλου ιδιαίτερου. Θα τα ανέφεραν ήδη οι διάφοροι ευρωβουλευτέ, τη σημασία τη πρόληψη. Στην προκαταρτική μελέτη για το πώς αγαπητοί μέλη υλοποίησαν την οδηγία, είδαμε ότι η πρόληψη είναι κάτι τα οποία έχουν πολλέ αδυναμίες στα κρατημέλη και απαιτείται ιδιαίτερη στήριξη με τη μορφή ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Επίσης, η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση για τα παιδιά και τους γονείς είναι κρίσιμη σημασία και ιδίως η εκπαίδευση των ε, ε, υπαλλήλων και υπευθύνων που είναι σε επαφή με τα παιδιά καθημερινά, στην καθημερινή τους δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερο, ένα συγκεκριμένο μέτρο πρόληψης που τονίζεται σωστά και από το σχέδιο γνωμοδότησης, η σημασία υποχρεωτικού ελέγχου του ιστορικού για άτομα, πρόσωπα, που θα εργαστούν ή θα προσφερθούν ως εθελοντές σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με τα παιδιά. Ως προς αυτό η ανταλλαγή πληροφοριών για όσους έχουν ε, κάνει παραβιάσεις, αδικήματα, αξιόπινες πράξεις όλη την Ευρώπη που έχουν σχέση με παιδιά είναι σημαντικό. Πρέπει να διευκολύνουμε την ανταλλαγή πληροφοριών για αυτά τα θέματα. Τέλος, κάτι που συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο έκθεσης, η υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων για τους παρόχους υπηρεσιών του διαδικτύου για υλικό ε, παιδικής εκμετάλλευσης που μπορεί να διαπιστώσουν στα δίκτυα. Την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ παρουσία του Γενικού Διευθυντή του ε, ε, Διεθνούς Κέντρου για την Προστασία των Παιδιών από την κακοποίηση της ΕΠΑ είδαμε πόση δουλειά έχουν κάνει ε, για την πρόληψη της ανάπτυξης τέτοιου περιεχομένου. Ο οργανισμός αυτός βοηθά πολύ και τις ευρωπαϊκές χώρες όταν χρειάζεται με ομάδες ανακριτών και την προσφορά βοήθειας για τη δίωξη των δραστών. Αυτά από δική μα πλευρά. Ευχαριστούμε την κυρία Φερχάριν και την Επιτροπή σα για την σχετική ομοδότησή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και από πλευρά μου στη Σαμπίνε Φερχάγεν για την πολύ καλή εργασία και την πολύ καλή πρόταση. Θέλω να το τονίσω. Τόσο αυτό που είπε τόσο ο συναδελφός Μίχελ, όσο και η κυρία πως πρέπει να προσέξουμε και να τονίσουμε περισσότερο την τήρηση των διαδικασιών του κράτους δικαίου και να μην έχουμε υπονόμευσή τους. Και εδώ να μην κάνουμε τους παρόχους υπηρεσιών σε οι οποίοι θα επιβάλλουν το δικό τους δίκαιο. Αυτό αποκλείεται. Και η αρχή του να διαγράφονται και να μην αποκλείονται περιεχόμενα είναι κάτι για το οποίο έχουμε αγωνιστεί πολύ στο παρελθόν και πιστεύω πως να την συνεχίσουμε, να την τονίσουμε και πάλι θα ήταν πολύ καλό ώστε να μην δημιουργηθεί η εντύπωση πως εδώ από την πίσω πόρτα πάμε να περάσουμε την αρχή του αποκλεισμού. Θα ήταν καλό να το τονίσουμε αυτό σαφώς. Θα ήθελα να ξαναδώσω στη Ζαμπίνε τον λόγο σύντομα και να υποδείξω πως η προθεσμία για τροπολογίες είναι η 11η Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για τις ιδέες των συναδέλφων. Πιστεύω ότι το θέμα θα άξιζε μια πιο μακρά συζήτηση, αλλά πιστεύω επίσης πως είναι πολύ σημαντικό να καταστήσουμε σαφές και εδώ πως δεν πρόκειται απλά για μια έκθεση Πρωτοβουλία αλλά για μια έκθεση εφαρμογής δηλαδή για να δούμε τι, έγινε, τι απέγινε η νομοθεσία πώς εφαρμόστηκε έτσι ώστε να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε στα σημεία για τα οποία έχουμε εδώ στην Επιτροπή ξεκάθαρη προτεραιότητα όπως είναι η πρόληψη λιγότερο η διάσταση του ποινικού δικαίου και πιστεύω πως σημαντικό είναι επίσης όσον αφορά την παιδεία, την κατάρτιση, την εκπαίδευση, την ενημέρωση και τα σχετικά μέτρα για νέους και παιδιά και για το προσωπικό που ασχολείται με παιδιά και νέους πρέπει να εστιάσουμε στους τομείς αυτούς. Θα ήθελα μόνο να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο το φαινόμενο αυτό ή μάλλον το πρόβλημα αυτό της σεξουαλικής κακοποίησης και της απεικόνησής του στο διαδίκτυο κατά κύριο λόγο δεν είναι πρόβλημα των ανοιχτών ιστοσελίδων. Εκεί βρίσκεται λίγο υλικό παιδική Το περισσότερο είναι κρυμμένο πίσω από άλλες σελίδες σε κωδικοποιημένο υλικό και έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα εδώ. Επίσης κατά την ποινική δίωξη, επειδή πολλοί τομείς σε πολλούς τομείς δεν έχουν πρόσβαση οι αρχές ποινική δίωξης. Οπότε δεν μπορούν να διαπιστώσουν την τέλεση αξιόπινων πράξεων και εδώ λόγω των ε, ένομων τάξεων που έχουμε πολλές φορές είναι δεμένα τα χέρια μας. Γι' αυτό και το πρόβλημα χρήζει της διεθνούς συνεργασίας η οποία λειτουργεί σχετικά καλά. Αλλά το πρόβλημα είναι πώς με τις ένομες τάξεις μας μπορούμε να προσεγγίσουμε τους δράστες οι οποίοι φυσικά και δεν εφαρμόζουν τις αρχές του κράτους δικαίου. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στο διαδίκτυο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να θέσω την ιδέα κατά πόσον μπορούμε από κοινού με την Europol να κάνουμε μια μικρή ακρόαση όταν είναι και ο Σκότισος εδώ στο ορατό μέλλον να ακούσουμε και πάλι την επικαιρότητα στο θέμα αυτό. Πρόεδρος. Χαίρομαι πολύ για τη συνεργασία. Πιστεύω πως θα είναι γόνιμη και καλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ιδέα αυτή στο τέλος. Πιστεύω πως όντως θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, να κάνουμε εδώ μια συζήτηση με την Europol. Θα παρακαλούσα μόνο για την να μου δοθεί κάποια ευελιξία, ώστε ίσως να το χωρέσουμε κάπου όπου ίσως ταιριάζει και όχι τους επόμενους δύο μήνες επειδή πιστεύω δεν θα τα καταφέρουμε τότε αλλά μπορούμε να το έχουμε κατά νου ώστε κατά τη διάρκεια του έτους ίσως να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων επί μια μισή ώρα στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 11 Μαΐου, 6 το απόγευμα, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εισηγήτρια και τους Σκιώδης και τους εύχομαι καλή επιτυχία στην εργασία τους. Περνούμε στο τελευταίο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Είναι η εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης για την έκθεση είναι είναι για τον έλεγχο δαπανών και παρακολούθηση της οικονομικής αποδοτικότητας των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εγγύησης για την Νεολαία. Δεν πέρασε πολύ καιρό, αλλά πριν από δύο εβδομάδες είχαμε μια πολύ εκτενή και πολύ καλή έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου το οποίο εξέτασε πόσο αποδοτικές είναι οι εγγύσεις για την νεολαία και ποιες επιτυχίες ή και αποτυχίες έχει στα κράτη-μέλη και πιστεύω πως τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής με δεν με χαροποιούν ιδιαίτερα, δεν είναι ιδιαίτερα θετικά. Πιστεύω πως πρέπει να εργαστούμε λίγο εντατικότερα έτσι ώστε οι εγγυήσει για την νεολαία να έχουν τις, τα αποτελέσματα που θέλουμε θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην Τερέζα Κομοντίνη, την εισηγήτρια. Παρακαλώ, συντομεύστε. Σε κάθε περίπτωση, όχι περισσότερο από πέντε λεπτά. Ήδη υστερούμε σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα λόγω τη ψηφοφορία. Κυρία Κομοντίνη. Thank you, Madam Chair. In fact, uh, um, Θα ξεκινήσω εκεί που σταματήσατε εσείς στο Ευρωπαϊκό, ε, το Ελληνικό Συνέδριο έκανε μια αξιολόγηση για το κατά πόσον η εγγύηση για την νεολαία δίνουν αποτελέσματα και ε, το κατά πόσον η πρωτοβουλία για την ε, ανεργία των νέων βοηθούσε. Εξέτασε το Ελληνικό Συνέδριο αν τα κρατημέλια κάναν πρόοδο στην εφαρμογή ε, της πρωτοβουλίας αυτής και ε, το κατά πόσο εξασφαλίζεται η βιώσιμη ε, ένταξη των νέων στην αγορά εργασία, η οποία αποτελεί ακόμα πρόβλημα. Επίσης εξαρτάται από την ποιοτική εκπαίδευση. Σύμφωνα με τις συστάσεις, ε, τα βήματα τα οποία ελήφθησαν στο πλαίσιο της εγγύησης για την νεολαία θα πρέπει να συμβαδίζουν περισσότερο με τις ανάγκες αγοράς. Παρατηρεί το Αναλυτικό Συνέδριο ότι κανένα κράτος μέλος δεν έχει κάνει μια πλήρη ανάλυση των αδυναμιών και των ελλείψεων που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες. Ένα αποτελεσματικό ε, πρόγραμμα εγγύηση για την νεολαία χρειάζεται να το παρακολουθούμε αποτελεσματικά και τα κράτη-μέλη να υποβάλουν τακτικέ εκθέσει. Σύμφωνα με το ελεγκτικό Συνέδριο, δεν έχει γίνει καμία πλήρη ανάλυση όλων των εκθέσεων που έχουν υποβληθεί. Ε, μια επαρκή αξιολόγηση των δεξιοτήτων και μια καλή ε, καταγραφή των αναγκών της αγοράς είναι απαραίτητες. Επίσης θα πρέπει τα στοιχεία που δίδονται να είναι συγκρίσιμα. Γι' αυτό το λόγο στην έκθεσή μου υπογραμμίζω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να ε, κάνει πιο αυστηρούς τους κανόνες ε, για τις εκθέσεις των κρατών μελών και για τις αιτήσεις του και, και επίσης ε, να δημιουργήσει ένα σύστημα ε, παρακολούθησης της εκτέλεσης των προγραμμάτων. Χρειαζόμαστε μια προσέγγιση, ισχυρή προσέγγιση εταιρική σχέσης με τα με τις εταιρείες, ε, ε, ιδιωτικές εταιρείες παροχής ε, υπηρεσιών απασχόλησης με τα κατα... ιδρύματα κατάρτισης, εκπαίδευσης κλπ. Τέλος, είναι πολύ σημαντικές οι δεξιότητες, ψηφιακές δεξιότητες, γιατί είναι απαραίτητες για την ε, εποχή μας και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τις συμπεριλάβουν και να τους δώσουν έμφαση. Αυτά είναι τα βασικά σημεία τα οποία θέλω να ε, συμπεριλάβω στην έκθεσή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κομοντίνη για την παρουσίαση της έκθεσής σας. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους κοιόδες εισηγητές Βλέπω τουλάχιστον ένα είναι εδώ. Η κυρία Δάρδια Σαβάλ Ρουβιάλ. Έχετε το λόγο για ένα έως ένα μισή λεπτό. Ε, Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Σημεριζόμαστε την θέση της εισηγήτριας. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ε, παρά τα υπέρ και τα κατά ε, Τη εφαρμογή, το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να υποστηριχθεί ε, παρά τι έλλειψει και τι αδυναμίε στην εφαρμογή. Άργησαν τα, άργησαν τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν ε, την εφαρμογή του, αλλά η κατάσταση έχει επιταχυνθεί πλέον, παρόλο ότι πολλά έχουν να γίνουν. Το αναφέρει αυτό το ελεκτικό συνέδριο. Το ελεκτικό συνέδριο έχει συστάσει, προτάσει, ιδέε προ τα κράτη-μέλη που θα πρέπει να τι λάβουν υπόψη του. Αλλά θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστέ. Όταν άρχισαμε να μιλάμε για τι εγγύσει για την νεολαία, ε, οι μελέτες έλεγαν ότι χρειαζόμαστε 45-50 εκατομμύρια κατέτος για να έχει αυτή η πρωτοβουλία πραγματικότητα. Ε, ε, το, οι, τα πόροι που έχουν εγκριθεί όμως είναι πάρα πολύ μικρότεροι, το 1,8 περίπου, ε, οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε και πάρα πολλά πράγματα. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωρίζετε ότι μπλόκαρε την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου για να προσθεθούν 1,8 δις ευρώ ακόμα. Ε, οπότε θα παραμείνουμε τα ποσά που είχαμε. Είναι σημαντικό να αξιολογηθεί αυτή η πρόοδος που έχει γίνει ε, από πλευράς βιωσιμότητας και πλευράς ποιότητας των προτάσεων. Αυτό θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα για την αξιολόγηση του προγράμματος αυτού. Όχι μόνο ο αριθμός των ατόμων που έχουν καλυφθεί, αλλά και η ποιότητα των προτάσεων, καθώς επίσης και η βιωσιμότητα. Θα πρέπει να προσθεθούν και αυτοί οι δείκτες, έτσι ώστε να γνωρίζουμε αν τα χρήματα τα οποία έχουν δαπανηθεί ήταν μια πραγματική προσθέμενη αξία ή απλώς χρησιμοποιήθηκαν έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να σταματήσουν να χρηματοδοτούν άλλου τύπου προγράμματα απασχόλησης. Δηλαδή να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα ποσά είναι πρόσθετα και δεν υποκαθιστούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ από το ECR. Δεν είναι πια κανείς εδώ. Από το ALDE επίσης δεν είναι κάποιος. Ο συνάδελφος Σούντες από το Γκουε ή θέλεις να πεις κάτι εκ μέρους του Γκουε, εντάξει. Στους πράσινους έχω τον συνάδελφο Μαραγκάλ, ο σκιώδη ο οποίος επίσης δεν είναι πλέον εδώ. Χέλγα, εσύ Εντάξει, ούτε η κυρία Μπίλτ είναι εδώ. Περνούμε λοιπόν στη συζήτηση από τα μέλη. Παρακαλώ, συνάδελφο Σέντροβα, να είναι σύντομη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, τη συνάδελφο Κομοντίνη. Είναι πολύ χρήσιμο το πρόγραμμα, όντω. Το πρόγραμμα λειτουργεί καλά, αλλά πρέπει να δώσουμε έμφαση στη διάσταση της αποδοτικότητας, τη γνωμοδότηση της εισηγήτριας. Σημειώνεται η έλλειψη πληροφοριών Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ακριβέστερη αξιολόγηση της ε, αποτελεσματικότητα προ το κόστο για κάθε κράτο και τη σχετική υποβολή εκθέσεων. Από αυτήν την έννοια θα υποβάλω σχετικέ τροπολογίες. Αυτά όλα και όλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να τοποθετηθεί. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει τότε θα ήθελα να υποδείξω Α, ναι. Λυπούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει τελικά. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ το πολύ δύο λεπτά. Very much. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και για τη γνωδότηση που καλωσορίζουμε. Είναι πολύ χρήσιμη συμβολή. Και ευχαριστούμε και για τη συζήτηση που γίνεται σήμερα και εμείς μελετούμε την έκθεση που μας έστειλε το και, ε, τα οποία τα περιλάβαμε και στην έκθεσή μας από το 2014. Η έκθεση αυτή επικεντρώνεται σε μια διετία στοιχείων, 2014-2015. Υπ' αυτήν λοιπόν την έννοια, δεν μπορούμε να έχουμε καταληκτήριες παρατηρήσεις και έχουμε εντοπίσει τις ελλείψεις που υπάρχουν στα αρχικά έτη της υλοποίησης. Κάποιοι τονίζονται ότι πρέπει να υπάρξει και ένα χρονικό πλαίσιο. Αυτό δεν απαιτείται ιδιαίτερος για τις εγγύσεις της νεολαίας. Πρέπει κυρίως να προβλέψουμε αρχές διαχείρισης, αρχές ε, που θα ασχοληθούν με την πραγματική υλοποίηση, την πρακτική υλοποίηση του προγράμματος. Πάντως από την ανακοίνωσή της του Οκτωβρίου η Επιτροπή λέει ότι η πρόσληψη της εγγύησης για τους νέους, ιδίως ως προς τη διάσταση των ΕΑΕΚ, ήταν πολύ επιτυχημένη. 16 εκατομμύρια νέοι ε, πήραν μέρος ήδη από πέρσι και άλλα πολλά εκατομμύρια ε, ζήτησαν να συμμετάσχουν σε προγράμματα διαβίου κατάρτισης και τα σχετικά 1,6 εκατομμύρια στηρίχθηκαν από το πρόγραμμα εγγύησης για τους νέους, δηλαδή το χρηματοδοτικό σκέλος. Βεβαίως αυτά θα αποδώσουν καρπούς ήδη στην πράξη. Κάποια κάτι μέλη ετοιμάζουν τις σχετικές παρατηρήσεις με ε, ε, κύριους παραλήπτες ακριβώς τους υπεύθυνους για την εγγύηση των νέων και κάποια παραδείγματα η εγγύηση των νέων στην Κροατία λόγω χάρη επέτρεψε τη δημιουργία ένα νέο σύστημα εντοπισμού που επιτρέπει στις δημόσιες υπηρεσίες να πάνε να βρουν αυτοί τους νέους που είναι δικαιούχοι τρόπον τεινά του συστήματος. Στη Φιλανδία έχουν δημιουργήσει μια νέα θηρίδα που δίνει τις σχετικές οδηγίες με χρήσιμες υπηρεσίες για ανέργους ή τους ΑΕΚ κάτω των 30 στη Γαλλία. Συνολικά προγράμματα χρησιμοποιούνται για την πρόορη εγκατάλειψη του σχολείου και την προώθηση της εκπαίδευσης στα σχολεία με μια πολύ στοχευμένη προσέγγιση. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα των μέτρων που μπορεί να έχουμε και το πώς μπορεί να υπάρχει στοχευμένη στήριξη προς τους νέους στην πράξη. Με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να σας διακόψω. Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ναι, ναι, πολύ γρήγορα. Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, Πρέπει να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση βεβαίω ω προ την παρακολούθηση λόγου χάρη από τα βασικά ζητήματα που έχουν τεθεί. Συνεργαζόμαστε και την Επιτροπή Απασχόληση, τι Επιτροπέ Απασχόληση των Κρατών Μελών, για να βελτιωθεί η παρακολούθηση και να έχουμε περισσότερα δεδομένα ω προ το κόστο, ω προ την ποιότητα των μέτρων σας ευχαριστώ πολύ για την γνωμοδότησή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που αναγκάστηκα να σας διακόψω με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι και ζήτημα δικαιοσύνης. Επειδή όταν διακόπτω τα μέλη της Επιτροπής, επειδή μακρηγορούν, πρέπει να κάνω το ίδιο και με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω πως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα είμαστε καταδικασμένοι να επιτύχουμε σε κάποιο βαθμό και σε αυτό το κοινοβούλιο πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε οι εγγύσεις για την νεολαία να γίνουν επιτυχία. Επειδή αν δεν μπορέσουμε να περάσουμε το μήνυμα στους νέους στην Ευρώπη πως έχουν προοπτική στη ζωή τους, τότε δεν μπορούμε να προσμένουμε από αυτούς να βλέπουν, να θεωρούν την Ευρώπη ως δική τους προοπτική. Γι' αυτό και πιστεύω πως είμαστε καταδικασμένοι να επιτύχουμε και πρέπει να κάνουμε τα πάντα η πρωτοβουλία αυτή να γίνει όντω επιτυχία. Γι' αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ την εισηγήτρια και θα ήθελα να τη δώσω ξανά σύντομα το λόγο υποδεικνύοντας πως η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η 7η Μαΐου στις 1 το απόγευμα. Η κυρία Κομοντίνη, εντάξει, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή εργασία στους στον, στους εισηγητές και τους κοιόδης. Φτάσαμε στο τέλος της συνεδρίασης και θα ήθελα να υποδείξω πως η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 29 Μαΐου από τις 3 έως τις 6.30 το απόγευμα και στις 30 Μαΐου από τις 9 στις 12.30. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ επίσης τους διερμηνείς οι οποίοι διευκόλυναν πάρα πολύ την εργασία μας όπως πάντα. αυτό και τώρα σας παρακαλώ εγκαταλείψτε γρήγορα την αίθουσα εκτός από τους συντονιστές και όλους αυτούς που πρέπει να συμμετάσχουν στο συντονισμό έτσι ώστε να μπορέσουμε γρήγορα να συνεχίσουμε την εργασία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή σας μέρα. Ich würde gerne mit der Koordinatorensitzung beginnen. I would like to... Θα ήθελα να αρχίσω με τη συνεδρίαση των συντονιστών τώρα. Επειδή ήδη έχουμε αργήσει λίγο,